πάντοτε στην παραγωγή την, ε, χωρίς να, να δίνουμε καλύτερη θέση στην ε, εργασία και την απασχόληση. E, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο